Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τανζάν πρέπει να σας πω ότι δεν θα είναι εδώ σήμερα. Είχε κάποιο ειδικό πρόβλημα, κάποια υποχρέωση ανηλυμένη και ήταν αδύνατον να έρθει σήμερα εδώ μαζί μας. Σύμφωνα με το γλασικό καθεστώς, ε, ξέρετε ποιες γλώσσες έχουμε, δανέζικα, φιλανδικά, λατινικά, βουλγαρικά, τσεχικά και στονικά δεν καλύπτονται. Να σας θυμίσω και τις διαδικασίες. Έχουμε ε, μετάφραση στις γλώσσες των τακτικών μελών που έχουν την προτεραιότητα ε, για τη διερμηνία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας. Επίσης μεταδίδεται μέσω διαδικτύου η συνεδρίασή μας. Είχαμε προβλέψει διευρυμένο προεδρείο στο τέλος της συνεδρίασης αυτής. Τελικά θα λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Αν έχετε παρατηρήσεις, τώρα παρακαλώ. Αλλιώς θεωρώ ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Έχω τώρα και κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω. Σύμφωνα με τον κανονισμό, άρθρο 192 παράγραφος 2, η Υποεπιτροπή αναθέτει στους συντονιστές κάποιες αποφάσεις για τη λειτουργία της, εκτός από την ψηφοφορία εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων και τροπολογιών, που προς το παρόν ε, παραμένουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο, στο οποίο κατέληξαν οι πρόεδροι ε, των πολιτικών ομάδων. 9 Νοεμβρίου σήμερα θα έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση. Έχουμε, θα έχουμε εδώ και τον κύριο Λαμαρά, ο είναι από την ε, ε, Αφρικανική Ένωση και θα έχουμε και το συντονιστή για την Αφρική από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Στεφιάτς επίσης θα είναι μαζί μας. Ο κύριος Λόπες Μπλάνκο που είναι διευθυντής για την Δυτική ε, Αφρική, επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης και τον κύριο Κέρχοφ επίσης, ο οποίος είναι συντονιστής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Έχουμε επίση και τον κύριο Θό. Στις 29 του μηνός είχα μια ακρόαση για το δικαίωμα τους συναθρίζεστε στο στρατό και έχουμε, είχαμε την ευκαιρία να καλέσουμε όλους όσοι ενδιαφέρονταν για το θέμα αυτό. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αυτής επίσης, θα θεωρηθούν τα πρακτικά εγκεκριμένα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα καλωσορίσουμε εδώ τον αναπληρωτή βοηθό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρίτσαρτ Φρό. Όπως γνωρίζετε, πριν από 10 μέρες έληξε η δράση του ΝΑΤΟ στη Λιβύη, Unified Protector, βάσει του ψηφίσματος 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να προστατεύονται οι άμαχος πληθυσμός και οι πολίτες της Λιβύης από τα στρατά του Καντάφη. Είπαμε και ακούσαμε εκεί τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από την επιτυχία αυτή η αποστολή, τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά όσο και τους στόχους που είχαν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Τα μαθήματα αυτά σίγουρα ε, θα συζητηθούν και στην επόμενη διάσκεψη που θα γίνει το Μέο του 2012 στο Σικάγο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη δικιά του την πλευρά παρακολούθησε τις εξελίξεις και τα γεγονότα στη Λιβύη από κοντά. Ο κύριος Μπούτζεκ, ο πρόεδρός μας, πήγε πριν από λίγες μέρες μάλιστα στη Λιβύη με μια ad hoc αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και ελπίζω ότι και εμείς θα επισκεφθούμε τη Λιβύη σύντομα. Τώρα επιπλέον από τα μαθήματα αυτά που μπορούμε να πάρουμε ε, από πολιτική και στρατιωτική άποψη έχουμε και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από αυτού θα ήθελα να έχω την άποψή σας για την σταθερότητα στη Λιβύη η κινητοποίηση επίσης και η ένταξη των μαχητών στην Νέα Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ, όπως επίσης και το θέμα της διάδοσης των ε, όπλων, το manpad όπως ονομάζεται. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και την ε, ε, πολιτική αεροπορία εφόσον ε, πέσουν ε, όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός στα χέρια αυτών που δεν θα έπρεπε. Γι' αυτό και εξετάζεται μία έκθεση όσον αφορά την κρίση που, τη δημοσιονομική κρίση και τον αντίκτυπό της στον αμυντικό εξοπλισμό. Είναι η έκθεση Λίζεκ. Επίσης εξετάζουμε το θέμα της ευρωπαϊκής ε, ε, ικανότητας, κάτι το αντίστοιχο με τις δυνάμεις ΜΑΡ του ΝΑΤΟ. Δεν θα σας εκπλήξει να ακούσετε πόσο πολύ μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, όπως επίσης και πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των όπλων ή και των δυσκολιών όσον αφορά την επιχειρησιακή ικανότητα της δράσης Unified Protector. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που σας έχουμε εδώ, κύριε Αναπληρωτή Βοηθό Γενικού Γραμματέα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ <clears throat> κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ενημερώσω περί της Λιβύης. Ε, πριν από αρκετές εβδομάδες μου είχε, ε, ε, μου είχε ζητηθεί να παρουσιάσω αυτή την ομιλία και συνεχιζόταν ακόμη η, η επιχείρηση προστασίας των πολιτών και ακόμη ακόμη ίσχυε το καθεστώς Καντάφη ενώ σήμερα η Λιβύη είναι ελεύθερη, έχει τελειώσει η περίοδος αυτή. Το προσωρινό Εθνικό Συμβούλιο ετοιμάζει μία μεταβατική κυβέρνηση και οι εξελίξεις είναι όπως τις παρουσίασε η Πρόεδρος. Έχει ξεκινήσει η μεταβατική περίοδος η οποία βέβαια παρουσιάζει προβλήματα και θα σας τα αναφέρω σε λίγο. Αλλά ελπίζω ελπίζουμε ότι η Λιβύη θα μπορέσει να καταλήξει σε μια διαδικασία ανοικοδόμησης και συμφιλίωσης και τώρα πρέπει ίσως να σκεφτούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις και αντιδράσεις της, Ευρω... της διεθνούς κοινότητος προς τη Λιβύη. Να σας πω πώς καταλήξαμε στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ για την ενοποιημένη προστασία και αυτή τη μοναδική επιχείρησή μας ε, με ε, διάφορους εταίρους συμπεριλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βεβαίως ε, η κατάσταση επιτόπου ε, και η ε, επέμβαση επιτόπου στη Λιβύη ε, πέτρεψε να εφαρμόσουμε πάρα πολύ γρήγορα και με τρόπο πρωτοφανή τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ και συγχρόνως να εφαρμοστούν τα μέτρα για να σταματήσει το καθεστώς Καντάφη τις εγκληματικές του ενέργειες βάσει των ψηφισμάτων του, της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ που επέτρεπε να χρησιμοποιήσουμε όλους τους αναγκαίους τρόπους για να προστατεύσουμε ε, τους πολίτες. Ε, γι' αυτό και πρόκειται για μια ιστορική εξουσιοδότηση. Στην αρχή της κρίσεως είχαμε καταρτήσει τρία βασικά κριτήρια. Πρώτον, μια σωστή νομική βάση, δεύτερον περιφερειακή στήριξη και τρίτον ε, ε, ε, κάλυψη όλων των αναγκών και ε, οι κινήσεις μας κάλυπταν και τα τρία κριτήρια γι' αυτό και στη συνέχεια ε, συζητήσαμε συχνά με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες και τους υπόλοιπους εταίρους μας για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε τις αναγκαίες δραστηριότητες με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητος πριν ακόμη εφαρμοστεί το ψήφισμα είχαμε προβλέψει την βοήθεια η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει κατόπιν ετήσεως ε, τη ΟΗΕ ε, και δύο ακόμη δυνατότητες τις οποίες ε, εφαρμόσαμε μαζί με την προστασία των πολιτών. Υπήρχε στενή συνεργασία μεταξύ του Γενικού Γραμματέα μας και της ΥΠΑ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, και ε, σε όλα τα επίπεδα, επίπεδο προσωπικού ή επίπεδο συμβουλίου μέχρι τη στιγμή της επεμβάσεως και ε, είχαμε εκπονήσει και σενάρια για την περίοδο μετά τον Καντάφη. Είδαμε λοιπόν ότι πολλές χώρες επενέβησαν άμεσα σαν δωρητές και μετά το ΝΑΤΟ ανέλαβε σαν συντονιστής για να υπάρχει ενοποιημένη προστασία και η επιχείρηση αυτή της ενοποιημένης προστασίας απέβλεπε σε τρία μέτρα. Καλυφθήκαμε με ε, αεροπλάνα, με ε, σε μια πολύ ευρεία περιοχή ε, όπου συμμετείχαν και τρεις χώρες που δεν συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ το Κατάρ, η Ορδανία, το Μαρόκο, η Σουηδία και ε, οι χώρες αυτές μπόρεσαν να στηρίξουν περιφερειακά τις ενέργειές μας. Η στρατηγική μας καθορίστηκε από την πολύ δύσκολη αποστολή μας να αποφύγουμε τις επιθέσεις κατά των πολιτών, πράγμα το οποίο σήμαινε ότι έπρεπε να εμποδίσουμε τους καταφικούς να ε, επιτίθενται με τάγκ και βαρύ πυροβολικό στο λαό της Βενγάζης αλλά και στη Μίστρα είχαμε ε, επέμβει ε, για να, ε, μπορούν, να μην μπορεί το καθεστώς να συντονίσει τις ενέργειές του είχαμε λοιπόν πάρα πολλές επιθέσεις από αέρα και πολλές επεμβάσεις σε πλοία ε, και πολλά από αυτά δεν επετράπει να προσεγγίσουν σε λιμάνι της επιλογής τους στη Λιβύη ε, ε, και καταστρέψαμε πάνω από 600 στόχους στην, επί του εδάφους ε, στηρίξαμε την ανθρωπιστική βοήθεια και μπορέσαμε να ε, εμποδίσουμε διάφορες κινήσεις για να ε, μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι αποστολές μας. Το ΝΑΤΟ δηλαδή ε, προχώρησε όπως απαιτούσαν οι ε, προϋποθέσεις που είχαν καταρτιστεί από το ψήφισμα. Είχαμε όμως δύο περιορισμούς. Ποτέ ε, δεν υπήρξαν υπό την καθοδήγηση του ΝΑΤΟ στρατεύματα ξηρά στη Λιβύη. δαπά και ήμασταν πολύ ακριβείς ε, ε, χρησιμοποιώντας ε, βλήματα μεγάλης ακριβίας και δεν έχουμε καμία επιβεβαιωμένη κατηγορία για θύματα επί του εδάφους παρόλο που είμαστε έτοιμοι να τεκμηριώσουμε τις απόψεις μας ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν μας Θέλαμε επίσης ε, μετά την ε, διαμάχη να αποκαταστήσουμε τη Λιβύη ως το δυνατόν πιο γρήγορα γι' αυτό και ποτέ δεν ε, είχαμε σαν στόχο το σύστημα ίδρευσης ή ηλεκτρισμού κατά τρόπον ώστε απλώς το καθεστώς να μην μπορεί να συνεχίσει την καταστροφική του λειτουργία και ποτέ δεν είχαμε σαν στόχο άτομα ακόμη και τον Καντάφη ε, και γενικώ πρέπει να πούμε ότι ήμασταν πολύ επιτυχημένοι και μπορέσαμε να περισσώσουμε χιλιάδες ζωές ακολουθήσαμε κατά γράμμα τις επιταγές που είχαν ε, ανατεθεί στο ΝΑΤΟ και εξασφαλίσαμε ότι η εργασία έγινε σωστά ε, η ε, επιχείρησή μας τελείωσε στις ε, ε, 25 Οκτωβρίου και ε, υπήρχε πλέον επαρκής σταθερότητα με, το, ε, με την Εθνική Μεταβατική Κυβέρνηση και το Συμβούλιο Ασφαλείας ανέλαβε μία παράλληλη ενέργεια και με το νεότερο ψήφισμα ανακάλεσε όλες τις εντολές οι οποίες είχαν δοθεί ε, μέσω του ψηφίσματος ψηφίσματος για την απαγόρευση υπερπτήσεων από τη Λιβύη και ε, για την επέμβαση. Ακόμη η υπάρχουν όμως διατάξεις οι οποίες ε, αναφέρονται σε ε, ένοπλη επέμβαση και μπορούν να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη ενδεχομένως. Ε, υπήρξε μία στήριξη στα μέτρα αυτά προς την Λιβύη και αποκομίσαμε και διάφορα διδάγματα για το ΝΑΤΟ ότι μπορούμε γρήγορα να καταρτήσουμε μία περίπλοκη ε, δράση εάν χρειάζεται χρησιμοποιώντας ηλεγμένα ε, προγράμματα και υπήρχε η Βούλη να ολοκληρωθεί ε, το έργο μας και η, προστα... Ε, ε, επιχείρηση αυτή απέδειξε ότι υπάρχει ένας ισχυρός πυλώνας του ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στηρίχθηκε και από τους Αμερικανούς ομολόγους και από τον Καναδά. Συγχρόνως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ γνώριζαν ότι υπήρξαν και ατέλειες σε πολλούς τομείς όπως η παρακολούθηση, η, ε, ε, ο ανεφοδιασμός με καύσιμα και θελήσαμε ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ατέλειες να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της εντολής του ΟΗΕ και ε, ε, ε, υπήρξε υπήρξε μια συντονισμένη κίνηση όλων των εμπλεκομένων για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Λιβύης και είμαστε έτοιμοι να συντονίσουμε ενέργειες σε οποιαδήποτε περίοδο μετά από μια κρίση η επιχείρηση αυτή και η πτώση του καθεστώτος του Καντάφη άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διότι πλέον μία χώρα μπορεί να ανανεωθεί, να υπάρξει εθνική συμφιλίωση η οποία μόλις αρχίζει και βεβαίως πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο λιβικός λαός θα, πρέπει να αναλάβει αυτή την ενέργεια και προς το παρόν υπάρχει ένα μεταβατικό συμβούλιο το οποίο πρέπει να καταρτήσει ένα κατάλογο προτεραιοτήτων των αναγκών του και μετά να ζητήσει βοήθεια από έξω. <clears throat> Υπάρχουν πρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και το πιο άμεσο αναφέρθηκε εις το τελευταίο ψήφισμα 2027 το οποίο αναφέρεται στον παρεμποδισμό της επεκτάσεως χρήσεως των όπλων όπου ζητείται να υπάρξει εξασφάλιση των συνόρων και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα καταρρεύσει το κράτος ε, ε, δικαίου και η ένομη τάξη. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε εάν μας ζητηθεί η βοήθειά μας αλλά δεν προσπαθούμε να βρούμε νέα καθήκοντα στη Λιβύη, Λιβύη ό,τι μας προταθεί θα εξεταστεί πολύ προσεκτικά και θα πρέπει να στηρίζεται από συλλογική ενέργεια και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε έναν πραγματικά νέο ο επαγγελματικό στρατό στη χώρα και αστυνομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης μπορεί να εμπλακεί αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε να υπάρχει το προσωπικό εγκαίρος και να στηριχθεί καθ' όλη την περίοδο ε, διότι έχουμε ενδιαφέρον να υπάρξει μια ανανεωμένη Λιβύη και να έχουμε σταθερότητα εις ε, την ε, ε, νότια όχθη της Μεσογείου που είναι στην πόρτα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Thank you for... Uh, σας ευχαριστούμε για την εισήγησή σας και θα δώσω το λόγο στον συντονιστή. Hans Thank you, Madam Chair. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις στον κύριο Φω και να τον ευχαριστήσω για την ενδιαφέρουσα συμβολή του σε αυτή τη συζήτηση. Ως πολιτικός είμαι, της από την ομάδα ALDE των Φιλελευθέρων στο Ευρωκοινοβούλιο και θεωρώ πως αυτή η επιχείρηση ενωμένη προστάτες ήταν επιτυχής. <clears throat> Οδήγησε στην επικράτηση της ειρήνης. Αλλά ως διεθνής ε, νομικός Είμαι, έχω κάποιες ερωτήσεις. Η, εντολή αυτή και η διάρκεια της ε, πεκτάθηκε, παρατάθηκε. Αν δούμε τώρα τις αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που λειτουργήσαν ως οι αεροπορικές δυνάμεις των επαναστατών τότε. Εσείς μπορεί να πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Υπήρχαν κάποια στρατεύματα επιτόπου για να εντοπίσουν τους στόχους. Ίσως να μην ήταν υπό τις εντολές του, τις του ΝΑΤΟ, αλλά ήταν υπό τις διαταγές των κρατών μελών. Και αν δούμε και το κομβόι του Καντάφη, από ό,τι κατάλαβα, ε, αποτελείται και από ένα γαλλικό αεροσκάφο. Ήταν υπό τις διαταγές του ΝΑΤΟ ή υπό τις γαλλικές διαταγές. είναι γαλλική επιχείρηση. Και το ρωτώ αυτό γιατί παρά τα θετικά αποτελέσματα η ερώτησή μου αφορά το κατά πόσο ή όχι ε, η εντολή, η αρχική <clears throat> τραβήχτηκε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε και έπειτα παρατάθηκε, θα παραταθεί μάλλον η εντολή για ακόμα μισό χρόνο. Από ό,τι ακούγεται είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Ευχαριστούμε κύριε Γολτιέρη. Σας ευχαριστώ. Εγώ ε, είμαι της ίδιας άποψης με τους συναδέλφους. το, αυτό που είπατε ότι η επιχείρηση θα έπρεπε να θεωρηθεί επιτυχής, όχι μόνο διότι τελικά εκπλήρωσε την εντολή της και επέτρεψε την αλλαγή του καθεστώτος, αλλά και επειδή ο περιορισμός ε, της απουσίας ε, στρατευμάτων επιτόπου και η ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων θυμάτων επετεύθη με εξαιρετικό τρόπο. Ενώ επηρεάστηκε το αποτέλεσμα, η έκβαση ας πούμε των, ε, της μάχης. Ε, γιατί συχνά ακούμε για χειρουργικές ε, βομβιστικές ενέργειες και επιχειρήσεις, αλλά κάθε φορά δυσπιστούμε. Αυτή τη φορά ωστόσο φάνηκε πως όντως αποφεύθηκαν οι απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, έχουμε και κάποιες αμφιβολίες και ερωτήσεις όσον αφορά το δόγμα και τις κάποιες νομικές πτυχές, καθώς και το θέμα του κατά πόσο συγκεκριμένα λειτουργήσε η αλυσίδα της, ε, του επιτελείου, η αλυσίδα των ε, ε, Ε, των διαφόρων επιπέδων. Ε, τώρα, εδώ βλέπουμε ότι ισχύει το δόγμα η ευθύνη προστατεύει και είμαι ευχαριστημένο με την επικράτηση αυτού του δόγματος. Ταυτόχρονα όμω, πράγμα που δεν είναι απαραίτητο επίκριση κατά τη επιχείρηση, αλλά δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να επιμένουμε να θεωρούμε αυτή την επιχείρηση ότι μπίπτει σε αυτό το δόγμα ευθύνη για την προστασία. Ενώ είναι σαφές ότι σε κάποια φάση μετατράπηκε σε κάτι διαφορετικό. Μετατράπηκε σε ένα είδος στήριξη σε μια εσωτερική διαμάχη που προσέφερε σημαντική στήριξη στους επαναστάτες, βοηθώντας τους να καταλάβουν την εξουσία. Και διερωτώ με λοιπόν από άποψη στρατηγική και δογματική, εσείς πώς μπορείτε να διορίσετε ε, αυτό που έγινε. Ποιος, πιο κοντά είναι στο τι έγινε στη Σερβία και στο Κωσιοπέδιο, αλλά και διαφορετικό επίσης, γιατί δεν υπήρχε επιτόπου, ε, δεν υπήρξαν επιτόπου επί, ε, επί ξηράς επιχειρήσεις. Έπειτα, όσον αφορά την αλυσίδα την επιτελική. Συχνά ακούσαμε ότι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ε, δικούνταν από μεμονωμένα κράτη, δηλαδή ε, επιχειρήσεις αεροπορικές που περνούσαν από συγκεκριμένο επιτελείο κρατικό όμως. Ε, όλοι περνούσαν μέσα από την ίδια επιτελική αλυσίδα ή υπήρχαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις που ήταν ε, ευθύνη των εθνικών επιτελείων. Πώς λειτουργήσαν όλα αυτά συγκεκριμένα και έπειτα ποιο ήταν το είδος της υποστήριξης που δόθηκε στα στρατεύματα των επαναστατών. δηλαδή, το ΝΑΤΟ δεν έπαιξε κάποιο ρόλο. Ναι, δεν είχαμε στρατεύματα επί τόπου στην ξηρά, δεν είχαμε στρατεύματα ξηράς, αλλά υπήρχαν κάποια στρατεύματα που εντόπιζαν στόχους ή έδιναν πληροφορίες για τις κινήσεις ε, των ε, στρατευμάτων. Ε, ακούσαμε και για κάποιες επιχειρήσεις συγκαλυμμένες. Το ΝΑΤΟ εδώ τι ρόλο έπαιξε, ήταν ευθύνη του ΝΑΤΟ ή ευθύνη των κρατών. Βέβαια καταλαβαίνω ότι μπορεί να μας πείτε και τίποτα είναι και δεν είναι και το των θυρών η συνεδρίασή μας, αλλά εμάς θα... για εμά θα ήταν ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι ακριβώς συνέβη. Και ο συνάδελφος ανέφερε το βαρδισμό του κομβόη του Καντάφη. Τελευταία μου ερώτηση αφορά αυτό που είπατε σε σχέση με τους περιορισμούς των ικανοτήτων, των δυνατοτήτων μας. Ε, και τον εντοπισμό αυτών. Για μας, ε, ως πολιτικούς, που σκεφτόμαστε τα διδάγματα των επιχειρήσεων της Λιβύης για την δικιά μας ε, πολιτική άμυνας, θα θέλαμε να ξέρουμε πιο συγκεκριμένα Πού βλέπετε μετά από αυτή την επιχείρηση να υστερεί η Ευρώπη ως Ευρώπη μετά την κρίση της Λιβύης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος Χριστόφ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Πολωνικά. Ο συνάδελφος Βολτιέρη είπε και ρώτησε ακριβώς αυτό που ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Οπότε, θέλω κι εγώ την απάντησή σας για αυτά, αλλά και κάτι ακόμα. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι στρατιωτικοί πυρογνώμονες είπαν ότι η επιχείρηση ε, πρόκειται να κρατήσει δύο ή τρεις μήνες παραπάνω. Αν μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι τόσο ισχυρή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχει στρατιωτικές ε, ικανότητες μεγάλες, αν ε, λοιπόν ισχύει αυτό, πιστεύω ότι ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο θα δυσκολευτεί να προσφέρει τους πόρους και ό,τι άλλο χρειάζεται, εξοπλισμό, ε, πυράβλους και τα λοιπά για να παραταθεί η επιχείρηση αυτή. Οπότε ρωτάω το εξής. Το ΝΑΤΟ ήταν προετοιμασμένο να συνεχίσει την επιχείρηση αυτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και όντως σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπήρχαν προβλήματα με στρατιωτικό υλικό, με πόρους, Οπότε να μην είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει κάτι με αυτά που ρώτησε και ο Ιταλός συνάδελφος και που έχει να κάνει και με τις συζητήσεις που γίνονται στη δικιά μας υποεπιτροπή εδώ και καιρό. Πρόκειται για την στρατιωτική ικανότητα γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολό της. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Η στρατιωτική ικανότητα των ε, κρατών μελών μέσα στο ΝΑΤΟ ρωτάω, μπορείτε εσείς να φανταστείτε μια τέτοια επιχείρηση σαν και αυτή στη Λιβύη να την κάνατε χωρίς τις Ηνωμένε Πολιτείε, μόνο δηλαδή με τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήταν εφικτό κάτι τέτοιο προς το παρόν, χρησιμοποιώντας μόνο την στρατιωτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μας χρειάζεται έτσι και αλλιώς η βοήθεια των συμμάχων μας και κυρίως των ΗΠΑ. Πρόεδρος, ωραία, και εγώ έχω να ρωτήσω μερικά πράγματα από την επιτυχή βέβαια αυτή η επιχείρηση ε, πήραμε αρκετά διδάγματα, κυρίως εμείς οι Ευρωπαίοι. Το πρώτο είναι ότι είμαστε ευάλωτοι, προκειμένου να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, γιατί τελικά το ΝΑΤΟ ανέλαβε το μεγάλο μέρος, αλλά ακόμα και σημαντικές χώρες, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, συμμετείχαν, ενώ άλλοι δεν μπόρεσαν να κρατηθούν πολύ στην επιχείρηση αυτή. Είναι ε, μια πραγματικότητα που μας κάνει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και θα ήταν καλό να εντοπίσουμε πού ακριβώς μπορούμε καλύτερα να συνεργαστούμε, να εντοπίσουμε δηλαδή αυτούς τους τομείς όπου μπορούμε όντως με τη συνεργασία μας να προσφέρουμε πολλά. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο έχει να κάνει με τις πληροφορίες, με την υπηρεσία πληροφοριών. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνεργασία και σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Και τέλος, για το μέλλον. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το μέλλον. Για μας τους πολιτικούς είναι σημαντικά αυτά που συμβαίνουν βέβαια σήμερα, αλλά είναι και σημαντικά αυτά που θα ε, συμβούν στο μέλλον στη Λιβύη. Ποιο είναι το μέλλον της Λιβύης όσον αφορά τα όπλα. Οι λιβικές αρχές έχουν αποδυναμωθεί τώρα όσον αφορά τον εξοπλισμό τους και δεν ξέρω αν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν όλες τις μελλοντικέ απειλές που θα τους έρθουν. Εσείς Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τις λιβικές αρχές ώστε να αποφύγουν άλλα μικρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το στρατιωτικό εξοπλισμό. Ευχαριστώ. Πολλές είναι οι ερωτήσεις σας. Θα τις απαντήσω ομαδοποιημένα για την ε, εντολή και τη διάρκεια της. Ήταν σαφής. Το Συμβούλιο ήταν ε, πολύ συγκεκριμένο. 28 ή 5, έτσι, ήταν και 5 μαζί, μην το ξεχνάμε. Αυτό κάθε φορά που συζητάγαμε για τη Λιβύη. Υπήρξε μια αλλαγή, θα θυμόσαστε, το Μάρτιο που ήταν το UNCR, είχαμε την ε, επιχείρηση που ξεκίνησε ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία μετά ανέλαβε τον ΝΑΤΟ και σιγά σιγά καταλάβαμε τον Απρίλιο ότι είχαμε πρώτον το G8 και μετά είχαμε και τους υπουργούς εξωτερικών του ΝΑΤΟ που συνεδρίασαν στο Βερολίνο. Συνέβησαν λοιπόν αυτά τα δύο σημαντικά γεγονότα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών στη συνάντηση αυτή αντιλήφθηκαν, ακόμα και οι Ρώσοι, ότι η πραγματική απειλή για τους πολίτες ερχόταν από τις δυνάμεις που στήριζαν τον Καντάφη. Επιβεβαιώθηκε αυτό και στο Βερολίνο. Οι προσπάθειες λοιπόν επικεντρώνονταν περισσότερο πώς θα εμποδίσουμε τις δυνάμεις αυτές του Καντάφη να επιτίθενται στους πολίτες. Ο συντονισμός ε, λοιπόν ξεκίνησε μετά από αυτή την ημερομηνία με τις δυνάμεις που ε, αντιτίθενται στον Καντάφη. Αυτές οι δυνάμεις μέσω εθνικών δικτύων έδιναν πληροφορίες παίρναμε αυτές τις πληροφορίες. Και επιπλέον είχαμε και τον υπολογαγό Μπουσάρ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της επιχείρησης αυτής, ήρθε στις αρχές της εβδομάδας στο Συμβούλιο και είπε ότι ναι εντάξει δεν μπορούσε ε, βέβαια να πει περισσότερα αλλά αυτό που είχε τότε ήταν ε, συμβούλους ειδικού μια ομάδα φυσικά ήταν μια βαριά αεροπορική επιχείρηση και από θαλάσσης, χωρίς ε, στρατοξηράς, έτσι. Αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα τι κάνανε οι αντίπαλοι των Καντάφη δυνάμεις, αλλά και δυνάμεις του Κατάφη είναι ότι προσπαθούσαν να καταλάβουν, ήταν κατά κάποιο τρόπο κάτι σαν ε, πολεμικό παιχνίδι, να προβλέψουν τα επιχειρησιακά σχέδια του Καντάφη. Οπότε, αυτό που θέλαμε είναι να μπορέσουμε να εμποδίσουμε τις αεροπορικές δυνάμεις του Καντάφη και έτσι να μπορούμε εμείς να ελέγχουμε τον ενέριο χώρο. Όντως, ε, παίρναμε πληροφορίες για τις επιθέσεις που εκείνοι ετοιμάζανε και δικοί μας ε, οι πιλότοι ε, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιθέσεις, να μην τις αφήσουν να γίνουν. Όντως γνωρίζαμε αρκετά καλά που ήταν οι διάφορες δυνάμεις, που υπήρχε απειλή για τους αμάχους και έτσι μπορούσαμε να επιτεθούμε. Ε, βλέπαμε που υπήρχε μεγάλη μετακίνηση ε, οχημάτων, που και αυτό θα μπορούσε να οδηγούσε σε απειλή των αμάχων. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Στόχος, για παράδειγμα, που αποφασίστηκε μέσα στην εντολή, αλλά μετά, μιλώντας, τι καταλάβαμε. Καταλάβαμε ότι γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας εκεί στην πόλη, οπότε περιμέναμε να τελειώσει ο ποδοσφαιρικός αγώνας, ώστε να έχουν φύγει οι άμαχοι και ε, να μην υπάρχει σχεδόν καθόλου απειλή για τους αμάχους ή περιμέναμε για τις επιθέσεις μας να τελειώσουν τα σχολεία. Μερικές φορές οι δυνάμεις του Κατάφη, πολύ εφιός. τι έκαναν, φρόντισαν να συγκεντρώνονται δίπλα στα σχολεία, σε νοσοκομεία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς περιμέναμε, περιμέναμε να λήξει το σχολικό ωράριο για να μπορούμε να φέρουμε σε πέρα τις επιχειρήσεις μας με ακρίβεια χωρίς να προκαλούμε ε, ζημιές ή ε, επιθέσεις από τις οποίες να πλήγονται και άμαχοι. Οι περισσότερες χώρες είχαν το δικό τους ε, αεροπορικό εξοπλισμό, όπως και στο Κωσυφοπέδιο. Οι διάφορες χώρες ξέρανε πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία είχε να είναι ακριβής στις επιχειρήσεις τους. Και όντω τα όπλα που διαθέτουμε σήμερα είναι πολύ περισσότερο ακρίβεια από ό,τι ήταν κατά το παρελθόν. Γι' αυτό και δεν έχουμε ε, πολλές απώλειες ε, αμάχων. Σίγουρα ορισμένε χώρες δεν διαθέτουν αρκετά τέτοια όπλα ακρίβειας, αλλά γι' αυτό και υπάρχει ένας οργανισμός όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπου γνωρίζουμε που υπάρχουν τέτοια όπλα τα μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Και ορισμένες χώρες που προσφέρουν, που σέπεθεραν δυνάμεις είχαν κάποια τέτοια όπλα και τα ε, μοιράστηκαν ε, με άλλους οι οποίοι έφεραν σε πέρα σε αεροπορικές αποστολές. Τώρα αν ήταν το ΝΑΤΟ ή αν ήταν σε εθνικό επίπεδο ήταν του ΝΑΤΟ η επιχείρηση. Το κάνουμε, το ΝΑΤΟ, έχουμε το σύστημά μας, το στρατηγείο μας, τη δικιά μας δίκηση Είχαμε λοιπόν στρατηγείο με υπηρεσία πληροφοριών που ενημερωνόταν, επεξεργαζόταν όλα τα δεδομένα που ερχόντουσαν από τα αεροσκάφη επανδρομένα ημί για να καθορίσουν τους στόχους. Και έπρεπε όμως να είναι σίγουροι, όχι απλώς σίγουροι, πολύ σίγουροι για τους στόχους, ότι όντως πρόκειτο για στρατιωτικό στόχο, αυτό που θέλαμε να πλήξουμε, και λάμβαναν υπόψη και τον περίγυρο ε, του στόχου, δηλαδή τι υπάρχει γύρω από το στόχο. Τώρα, αν ε, υπήρχαν λήψεις από πλευράς Ευρώπης, κοιτάξτε, σίγουρα οι Ηνωμένε Πολιτείε βοήθησαν κυρίως με πληροφορίες. Αναλύσαμε τα πρώτα διδάγματα από αυτή την επιχείρηση. Οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί συμμαχοί έχουν κάποιες ικανότητες, αλλά όχι σε μέγεθο, σε αριθμό όπως και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό και οργανωνόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο και πρέπει κι άλλο να οργανωθούμε στο ΝΑΤΟ για να δούμε πώς θα έχουμε το εύρος εκείνων ικανοτήτων, επιχειρησιακών ικανοτήτων που θέλουμε να έχουμε και ίσως βάζοντας μαζί τα πυρομαχικά μας για παράδειγμα. Με πυρογνώμονες στο ΝΑΤΟ προσπαθούμε όντως να δούμε σε διεθνέ επίπεδο πώς μπορούμε να βάλουμε τις δυνάμεις μας μαζί και να μπορούν όλα τα αεροσκάφη να χρησιμοποιούν όλα τα πυρομαχικά για παράδειγμα και όχι να φτιάχνουν ορισμένα πυρομαχικά μόνο για ένα τύπο αεροσκαφών που να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Να υπάρχει διαλειτουργικότητα δηλαδή. Ένας άλλος τομέας είναι ο ανεφοδιασμός. Και εδώ στηριχτήκαμε πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ανεφοδιασμό. με τα αεροπλάνα πας, φέρεις επέρα στην αποστολή σου και επιστρέφεις. Είχαμε όμως όπως ξέρετε ε, βάσεις και στην Ελλάδα και στην Ιταλία που από εκεί πηγαίνανε στην Λιβύη, φέρασε σε πέρα στην αποστολή τους και επιστρέφανε. Είναι ένας περίπλοκος, ε, μια περίπλοκη χορογραφία θα έλεγα που έπρεπε να λάβει η χώρα γιατί πρέπει να προστατεύει συγχρόνως τα αεροσκάφη σου που πάνε, που πρέπει να πάνε στο συγκεκριμένο σημείο, που πρέπει η σειρά των ε, δραστηριοτήτων να λαμβάνει η χώρα ακριβώ όπω πρέπει. Δηλαδή, ποια στιγμή πρέπει να γίνει ο ανεφοδιασμό. Και χρειάζονται και πληροφορίε, βέβαια, οι κατάλληλε από τι υπηρεσίε πληροφοριών, οι οποίε πρέπει να είναι ακρίβειε και να ενημερώνονται συνεχώ. Ρωτάτε. Μάλλον ο ανέφερε, λέτε, πολύ το κατά πόσο οι Ευρωπαίοι στάθηκαν στο ύψος, είχαν ε, τις δυνατότητες να συμμετέχουν κτλ. Ναι, ναι, Φυσικά με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών που παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ανεκτήμητο. Η πραγματική πάντως επιχείρηση έγινε από τους Ευρωπαίους και τον Καναδά. Αν χρειάζονται περισσότερα, ναι. Και όλο αυτό το θέμα της Smart Defense και του να βάσουμε από κοινού τις δυνάμεις μας είναι ακριβώς για να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα με τα ίδια χρήματα σε καιρούς οικονομικής κρίσης όπως αυτής ο οποίος βρισκόμαστε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά πρέπει κάτι να βάζει κανείς για την άμυνα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε άμυνα χωρίς να ξοδεύουμε και ότι μπορούμε να την καταργήσουμε. Γιατί όταν θα τη χρειαστούμε δεν θα μας έρθει σαν το διακόπτη, το ανάβουμε ή τον σβήνουμε. Δεν γίνεται έτσι, πρέπει να το προετοιμάσουμε. Πρέπει να αναπτύξετε την άμυνά σας, να τη σχεδιάσετε, να εκπαιδεύετε. Άρα πρέπει να βάζουμε χρήματα στην άμυνα. Και πρέπει να κάνουμε καλύτερα πράγματα από ό,τι μέχρι τώρα. Και ένας τρόπος είναι το λεγόμενο pooling and sharing, δηλαδή να βάζουμε μαζί τις δυνάμεις μας, τους πόρους μας, ε, να έχουμε τις κατάλληλες συμβάσεις με την βιομηχανία, ώστε να έχουμε ό,τι μας χρειάζεται, να εναρμονίζουμε τις ε, απαιτήσει μας, να τις αναπτύσσουμε με τον ίδιο τρόπο και έτσι να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Και αυτό θα γίνεται εφόσον διαθέτουμε του ίδιου είδους εξοπλισμό όλοι. Οι πληροφορίες τώρα, η υπηρεσία πληροφοριών. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες. Δεν υπήρχε από την αρχή στο βαθμό που θέλαμε, αλλά όσο πέρναγε ο καιρό, ε, πήγαινε πολύ καλά. Όντω, οι πληροφορίες ερχόντουσαν, ε, οι πληροφορίες που χρειαζόντουσαν οι δυνάμει για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στις επιχειρήσεις τους και τι χρησιμοποιούσαμε όλο και περισσότερο. Υπήρχαν αρκετές πληροφορίες ώστε να πετύχουν ό,τι πέτυχαν οι δυνάμει μα. Να επιτύχουν δηλαδή. Τώρα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Η βοήθεια μπορεί να έρθει και από τις ε, κυβερνήσεις ε, για τις χώρες ε, αυτές της Βόρειας Αφρικής. Σε τόσο καιρό είχαν τα προβλήματα που είχαν. Μπορούμε να τις βοηθήσουμε προτείνοντας λύσεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και η διεθνής κοινότητα και όλες οι χώρες ξεχωριστά μεταξύ τους μπορούν να βοηθήσουν τη Λιβύη με τους θεσμούς της δίνοντας συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις, την αστυνομία τους, να έχουν ένα καλό δικαστικό σύστημα. Το καλό νέο με τη Λιβύη, ακριβώς επειδή δεν καταστράφηκαν πολλοί υποδομές, μπορούν ξανά να παράγουν πετρέλαιο, να προχωρήσουν σε εξόριξη πετρελαίου, να το πουλήσουν και έτσι να κερδίσουν πολλά χρήματα από τη διεθνή κοινότητα, η οποία πρέπει να τους βοηθήσει όμως χρειάζονται τη βοήθειά μας και τους τη δίνουμε ευχαρίστως. Thank Σας ευχαριστώ. Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, συνάδελφοι. Yeah. Thank you very much, uh, It's... Uh, Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φρό. Είναι πολύ ενδιαφέροντα το όσα μας είπατε. Εγώ έχω μια λεπτή ερώτηση, αν μπορείτε κάπως να επεκταθείτε. Ποιος θα τα πληρώνει όλα αυτά? Υπάρχουν, ε, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Υπήρχαν πολλά χρήματα δε της χώρας του Καντάφη παγωμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Εγώ παρακολούθησα πολύ στενά την κατάσταση και δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Ελπίζω πως θα βρεθεί κάποια συμβαστική λύση, γιατί μπορεί να υπάρξουν επιχειρήσεις σε χώρες όπου ο κόσμος δεν μπορεί να τα πληρώσει όλα αυτά. Θα ήταν καλό λοιπόν για το μέλλον να βρεθεί κάποια συμβαστική λύση. Ποια είναι η δική σας γνώμη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουτικόφερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην αρχή οι Κινέζοι και οι Ρώσοι απέχοντας ε, από το Συμβούλιο Ασφαλείας άνοιξαν το δρόμο για να γίνει αυτή η επιχείρηση, να υλοποιηθεί. Ε, μετά από λίγο άρχισαν να ερμηνεύουν την, να, μάλλον να επικρίνουν την ερμηνεία του ΝΑΤΟ πολύ έντονα. Στο τέλος οι Κινέζοι ήρθαν και περιέγραψαν τον Καντάφη ως εχθρό του λαού του, αλλά διερωτώ με αν είχατε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για το πώς αυτοί αξιολογούν την επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Θα τον ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Στην τελευταία συμφωνώ ότι θα ήταν ενδιαφέρον να είχαμε επαφή. Δεν είχαμε όμως με τους Κινέζους ακόμα. Αλλά έχετε δίκιο ότι υπήρξε μια αλλαγή στη διεθνή κοινότητα. Ότι πέρασε όντως αυτό λόγω της αποχής των Κινέζων και των ε, ε, Ρώσων, τα πρώτα δύο. Το, το τελευταίο, το 2009, ήταν ομόφωνη η απόφαση. Υπήρξε μετακίνηση στην κατανόηση του τι γινόταν καθώς περνούσε ο καιρός. Και νομίζω πως τελικά όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν και στήριξαν πλήρως τις ενέργειες που έγιναν και το ρόλο και το δρόμο μάλλον που ακολουθούσε η Λιβύη. Οι Κινέζοι δεν μας προσέγγισαν και ούτε και εμείς τους έχουμε προσεγγίσει. Μπορεί να υπάρξει κάποιο βήμα που θα γίνει σχετική συζήτηση και να προκύψουν οι απόψεις αυτές, αλλά θα δούμε. Το θέμα για το ποιος θα πληρώσει όλα αυτά. Φαντάζομαι ποιος θα πληρώσει για την επόμενη φάση εννοείται και τη στήριξη. Είμαι βέβαιος πως οι Λίβοι θα κάνουν τη δική τους συμβολή και αυτό είναι το πλονέκτημα αυτών των χρημάτων που ξεπάγωσαν, που θα το πάρουν δηλαδή τα χρήματα αυτά από τις πωλήσει του πετρελαίου. Ότι δηλαδή θα έχουν τα μέσα να ξαναχτίσουν τη χώρα τους, να φτιάξουν τους θεσμούς, να φτιάξουν την κυβέρνηση που χρειάζονται για να προχωρήσουν. Δεν, δεν νομίζω πως ζητήσατε να, να πληρώσουν για τη δική μας επιχείρηση. Δεν το κάναμε αυτό για να βγάλουμε λεφτά. Αυτό είναι προς το συμφέρον των ε, ε, κρατών του ΟΗΕ και της Ένωσης η Λιβύη να είναι μια σταθερή παραγωγική χώρα, μέλος της διεθνής κοινότητας. Ένα παραπάνω καθώ είναι στο κατόφλι μα, είναι γείτονε. Κάποια στιγμή θα βοηθήσουν και εκείνοι με τη σειρά του άλλου στην γειτονιά αυτή και θα είμαστε όλοι ισχυρότεροι. Ναι, με αυτό συμφωνώ μαζί σα απολύτω. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και υπήρχε με ένα προηγούμενο στο Κουβέιτ όταν μπήκε μέσα ο Σαντάμ και εκείνοι συνέβαλαν, είχαν αρκετά χρήματα και πλήρωσαν για αυτές τις επιχειρήσεις. Εμείς δεν τους ζητάμε τους, Λίβιου, Λίβιους, δεν είναι το ίδιο με, τους, ε, το Κουβέιτ, αλλά θα ήταν καλό ε, σαν συμβαστική λύση. Υπάρχει ένα σωρό χρήμα εκεί και η καιρή είναι δύσκολη για όλους. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι όχι, δεν το, κάνετε, δεν το κάνουμε για τα λεφτά, όχι βέβαια. Μάλιστα, υπάρχουν άλλε ερωτήσει. Όχι. I Θέλω να σα ευχαριστήσω για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Η παρουσίασή σας ήταν πραγματικά ανοιχτή και σημαντική για μας, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τι επιχειρήσει αυτές. Εμεί σε αυτήν την Επιτροπή Στηρίζουμε αυτή την αρχή. Όλες οι ερωτήσεις δείχνουν το ενδιαφέρον της ε, Επιτροπής για τη Λιβύη. Είναι η πρώτη επιχείρηση στη δική μας εντολή που μας δίνει την ε, δυνατότητα να αποκομίσουμε κάποια διδάγματα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω εξ ονόματος της Επιτροπής για την ε, καρποφόρα συνεργασία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. The next uh, on the agenda uh, Επόμενο θέμα της κυρίας διάταξης είναι η περίφημη έκθεση του κυρίου Λίσεκ. Σύμφωνα με τη διαδικασία θα δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Λίσεκ για να μας την παρουσιάσει. Έχετε το λόγο, Κρίστο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εσείς όχι μόνο προεδρεύετε λοιπόν εδώ, αλλά είστε και σκιώδη συζήτρια για την ομάδα ALDE. Έχουμε λοιπόν συζητήσει την έκθεση αυτή χτες. Δεν πιστεύω πως θα έχει νόημα να σας παρουσιάσω την έκθεση λεπτομερό σήμερα. Και πρέπει να συζητήσουμε τις τροπολογίες και τις συμβαστικές προτάσεις που έγιναν. Ένα σχόλιο μόνο που κατά τη γνώμη μου επιβεώνει την άποψη πως η... γενικά η έκθεση αυτή και η ουσία της είναι θετική και σωστή. Καθώς ακούω τον κύριο Φρόγα που, που δουλεύει για τον ΝΑΤΟ, είχα την αίσθηση ότι ήταν τελείως εκτός της ε, έκθεσης μου. Μίλησε για την ε, μοιρασιά των πόρων, για τον καλύτερο προγραμματισμό, για την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, όλα αυτά τα στοιχεία ε, περιλαμβάνονται και στην έκθεσή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους όσους ασχολήθηκαν και κοίταξαν την έκθεσή μου και καταρχήν τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά επίσης και άλλους συναδέλφους, διότι λάβαμε διάφορες τροπολογίες από διάφορους ε, βουλευτές και μέλη της Επιτροπής μας, της Υποεπιτροπής μας. Και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία Αυτόν βελτιώνει την έκθεσή μου και ότι συμφωνώ με τη μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών που έλαβα. Θα ήθελα μόνο να εξηγήσω γιατί κάποια από τα στοιχεία που αναφέρατε στις δικές σας τροπολογίες δεν, δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική εκδοχή της έκθεσης. Δεν ήθελα να επαναλάβω τις πολύτιμες δηλώσεις που είχαν συμπεριληφθεί στην έκθεση από τον κύριο Γκουαλτιέρη ή από τον κύριο Ντανζόν. Πρόσφατα ε, είχαμε ψηφίσει πάνω σε αυτές τις εκθέσεις και αυτά όλα είναι νοπά στη μνήμη μας και γι' αυτό δεν θέλω να τα επαναλάβω. Αν όμως αυτό είναι η βούληση της πλειοψηφίας, μπορούμε να περιλάβουμε αυτά τα στοιχεία στην έκθεσή μου. Για όσους δεν ήταν παρόντες στη χθεσινή συνεδρίαση, θα ήθελα να σας πω ότι καθώς συναντηθήκαμε με τους και οδησίγητες, Είχαμε μια πολύ καρποφόρα συνεδρίαση και τελικά επιτύχαμε συνεργασία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων και συμβαστικές λύσεις που εγώ είχα προτείνει στο 99% των περιπτώσεων ε, και νομίζω ότι το υπόλοιπο απλώς ε, θα είναι αντικείμενο συμβαστικών τις επόμενες μέρες. Μαζί με τους και ηγητές κυρία Κοπά και Νικολάη αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε άλλη μια συνεδρίαση στο Στρασβούργο την Τρίτη ε, για να έχουμε κάποιο χρόνο παραπάνω να το συζητήσουμε με τις πολιτικές μας ομάδες το θέμα. Αυτά λοιπόν εισαγωγικά και όπως σας είπα είμαι ανοιχτό για τα σχόλια και τις προτάσεις σας και με ευτυχής που βλέπω ότι τα σχόλια σας και οι προτάσεις σας εμπλουτίζουν την έκθεσή μου. Κύριε Κοπά. As Όπως ε, ήδη αναφέρατε θα χρειαστεί κάποια βελτίωση ε, στις λεπτομέρειες των ε, τροπολογιών αλλά τα βασικά έχουν συμφωνηθεί και νομίζω ότι είναι σαφές το μήνυμα ότι πρέπει να προωθήσουμε την περαιτέρω προώθηση της πολιτικής και ε, να υπάρχει μία συνεργασία για να εφαρμοστεί οι ρήτρε αλληλεγγύης ε, αυτής ε, αυτού του οργανισμού αμήνης. Δηλαδή, να δούμε Ε, τι μπορεί να γίνει διότι θεωρούμε ότι η προώθηση της βιομηχανικής βάσεως μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία βιωσίμων θέσεων εργασίας και βιομηχανιών με, το ελάχιστο, με την ελάχιστη ε, δυνατή επίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν να ε, βασιστούμε εις ε, την συμπληρωματικότητα και την αλληλεπίδραση κατά τρόπον ώστε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Είναι όμως επίσης βασικό να υπάρχει μια διαδικασία της οποίας θα ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ταμεία θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και υπέρ της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας. Σας υπενθυμίζω την τροπολογία μου 51 που υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες κατά τρόπον ώστε να προωθηθεί το θέμα και στην πολιτική γυτνιάσεως να υπάρξει ένα πολιτικό ε, μέσο πιέσεως ε, για βελτίωση της κατάστασης. Ο κύριος Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Λίσεκ για το σχέδιο εκθέσεως και για την εργασία την οποία έκανε στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Η κατάσταση είναι ακριβώς αυτή. Προσπάθησε να δημιουργήσει μία συνένεση και να την ε, ενσωματώσει και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Έχω όμως ορισμένες παρατηρήσεις εκ των οποίων δύο μπορούν να επιληθούν πιο εύκολα αλλά άλλες δύο ε, αντικρούν σε μεγάλες αντιρρήσεις. Καταρχήν ήθελα να αναφερθώ εις ε, τη συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 4 όπου στην αρχή λέγεται το εξής ε, Reiterate his views» επαναλαμβάνει την άποψη ότι μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή άμυνα θα βελτιώσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και ε, θα δώσει μια σημαντική συνδρομή στη συλλογική ασφάλεια στα, περιπλάσια, στα, στα πλαίσια του ΝΕΤΟ. Για μένα αυτή η φράση είναι αμφιλεγόμενη διότι ο, σαν στόχος η η στρατηγική αυτονομία αντικρούει εις το επόμενο κείμενο διότι στρατηγική αυτονομία και στο περιβάλλον του ΝΑΤΟ δεν συνάδουν διότι είναι σωστό να αναφερόμαστε εδώ στο ΝΑΤΟ αλλά στο παρελθόν βάσει της εκθέσεως Γκουαλτιέρη έχουμε χρησιμοποιήσει και συμφωνήσει μία άλλη γλώσσα και αναρωτιέμαι αν δεν μπορούμε να την επαναλάβουμε να μιλάμε για strategic relevance ή για strategic potential ή κάτι τέτοιο αλλά strategic autonomy ε, παρουσιάζει μία ε, ε, προοπτική την οποία δεν θεωρώ ότι είναι ούτε ρεαλιστική ούτε τότε ε, ε, πρέπει να την προσπαθήσουμε. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να προωθήσουμε το κείμενο ή στην συνέχεια, δηλαδή να λαμβάνουμε υπόψη μας στο ΝΑΤΟ και θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούμε να βρούμε μία άλλη διατύπωση. Το δεύτερο μου θέμα αναφέρεται στην παράγραφο 25 όπου μιλάμε για την Βαϊμάρη. Και εδώ ήθελα να ρωτήσω αν αυτό μπορούσε να ενισχυθεί κάπως, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής μεταξύ έχουμε προχωρήσει, έχουμε τη Βαϊμάρη συν, δηλαδή με την Ισπανία και την Πορτογαλία και την Ιταλία με συγχωρείτε λέει ο μιλητή σε κάποιο σχόλιο που δεν ήταν στο μικρόφωνο. Ε, θα μπορούσαμε όμως να συμπεριλάβουμε και τη Βαϊμάρη ε, Plus και να ενισχύσουμε τη διατύπωση αυτή. Αλλά τα δύο θέματα στα οποία αναφέρομαι ε, και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη αντίρρηση και που δεν είναι σωστή η κατεύθυνση είναι αφενός όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στην ε, στο μελλοντικό άνοιγμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για θέματα εξοπλισμών. Θεωρώ ότι αυτό είναι λανθασμένο. Υπάρχει ακόμη ε, μία εθνική πολιτική και επικάλυψη. Με το... Δεν πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε ε, ένα, μία επικάλυψη με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για τον οποίο ούτως ή άλλως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και δεν θεωρώ ότι είναι λογικό εάν προσπαθούμε να τον μειώσουμε να περιλαμβάνουμε ε, θέματα εξοπλισμών. Επίσης αν δούμε δούμε τι διεξάγεται ή στην ε, κοινωνία των πολιτών βλέπουμε από τα 141 ε, εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων έχουν αποδοθεί 93 σε προγράμματα τα περισσότερα δηλαδή το 75% έχουν αποδοθεί σε ένα πρόγραμμα στο ε, Τάλις και αντιλαμβάνεστε ότι και για τα στρατιωτικά διαφορετικά θα γινόταν το ίδιο αν τα αφήναμε να μπουν από την πλαϊνή πόρτα. Εάν λοιπόν θέλουμε ε, να ανοίξουμε την πόρτα πιστεύω ότι αυτό θα είναι μία λανθασμένη κίνηση και θα οδηγήσει ε, ότι μεγάλες επιχειρήσεις ε, όπως ε, η ΕΑΝΤΕΣ και το ΤΑΛΙΣ θα κυριαρχήσουν την αγορά, θα αρχίσουν να ροκανίζουν τον προϋπολογισμό μας και θεωρώ ότι αυτό είναι τελείως λανθασμένος. Δηλαδή οι παράγραφοι που αναφέρονται στα θέματα αυτά από 32 και μετά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να δεχτώ ε, ε, και πιστεύω ότι το 57 και 58 ε, να πληρώνουμε άλλα προγράμματα από τον εξοπλισμό αυτό δεν είναι σωστό από τον προϋπολογισμό αυτό δεν είναι σωστό και επίσης Θεωρώ ότι τα χρήματα μπορούν να ληφθούν από το εργαλείο σταθερότητα. Δηλαδή, εάν αφαιρέσουμε από εκεί χρήματα διαχειρίσεως κρίσεων για άλλα θέματα τα οποία προωθούν πολιτιστικά ανοίγματα, είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει και δεν μου φαίνεται εφικτό επιπλέον. Το δεύτερο θέμα και αναφέρομαι εδώ λιγότερο στον εισηγητή και περισσότερο σε, άλλους, σε θέματα που έχουν θέσει άλλοι συνάδελφοι ε, ε, πιστεύω ότι εδώ είναι σαν να μην είμαι στην Επιτροπή Υποεπιτροπή Ασφαλείας αλλά στην Επιτροπή Απασχόλησης. Η, η πολιτική αμήνης δεν είναι πολιτική απασχόλησης και δεν πρέπει να την ε, ε, χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή στο 12, 13, 14 όπου ζητάμε ε, να αγνοήσουμε την οδηγία για τις ευρωπαϊκές δημόσιες προμήθειες για την οποία έχουμε πολεμήσει επί χρόνια και άλλα δεν είναι δυνατόν να λέει το Κοινοβούλιο ότι κάνουμε πίσω σε πράγματα τα οποία ε, έχουμε προσπαθήσει. Αυτά. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι μεγάλες πρόεδροι και μπορώ να τα στηρίξω. Ε, μπορώ να μιλήσω για την Ρουμανία και να σας εξηγήσω την, ε, τα θέματα αυτά. Όσον αφορά την συνεργασία θα ήθελα να σας πω ότι οι φιλελεύθεροι συμφωνούν με το όραμα αυτής της εκθέσεως και στηρίζουν και ε, τις ε, τροπολογίες. Θεωρώ λοιπόν ότι η πολιτική αμήνης σε μια Ευρώπη σε κρίση, διότι αυτό εξετάζουμε στην έκθεση αυτή, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση και πόσο μπορούμε να εξασφαλίσουμε μία σωστή πολιτική αμήνη στα κράτη-μέλη διότι ελέγχθη ότι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία θα χρειαστεί να επιλύσουμε και ότι δεν έχουμε πάντοτε επαρκούς, επαρκείς πόρους για να το πετύχουμε. Πρέπει όμως να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μία βιομηχανία αμυντική που να είναι ισχυρή να βασίζεται στον ανταγωνισμό και συγχρόνως να λειτουργεί προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν ξέρω ε, αν οι ε, πόροι θα καταλήξουν στην ΕΑΝΤΕΕΦ ή σε άλλες επιχειρήσεις, αλλά θεωρούμε ότι ε, τα στοιχεία αυτά μπορούν να επιτρέψουν μία προστιθέμενη αξία προς την ευρωπαϊκή Αμερική αμυντική βιομηχανία. Επιπλέον πρέπει να προωθήσουμε αυτή τη βιομηχανία. Χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας και εις την αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αριστεριστές ή ότι θέλουμε να εμφανιστούμε σαν αριστεροί, απλώς θέλουμε να στηρίξουμε ορισμένα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Όλοι Όλο τον καιρό μιλάμε για την ε, μείωση ε, των δυνατοτήτων μας αμήνης και αυτό επηρεάζει την αμυντική μας πολιτική την οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ε, μία λύση για να παραμείνει ο εξοπλισμός μας τουλάχιστον στο ισχύον επίπεδο και θα πρέπει να προωθήσουμε την αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη και γι' αυτό συμφωνώ με τις συμβιβαστικές τροπολογίες όπως έχουν διαμορφωθεί και τις στηρίζουμε. Αυτή η έκθεση ουσιαστικά ακολουθεί ε, μία ε, παράδοση του κοινοβουλίου αυτού, δηλαδή συνοδεύεται από δηλώσεις, αλλά ε, θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή δεν έχει συζητηθεί από πλευράς κομματικών σκοπιμοτήτων και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τις ε, κομματικές σκοπιμότητες και ιδεολογίες αλλά να τις ξεπεράσουμε. Ε, υπάρχουν βέβαια συμβιβαστικές τροπολογίες ε, στις οποίες πρέπει να υπάρξει βελτίωση και θα τις συζητήσουμε στο Στρασβούργο αλλά πιστεύω ότι η έκθεση Λίζεκ είναι εξαιρετική για τον τομέα τον οποίο πραγματεύεται και θα την ακολουθήσουμε και σας ευχαριστώ. Κύριος Γουαλτιέρη. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, κάνετε καλή δουλειά. Ωστόσο, υπάρχουν ε, κάποια σημεία ακόμα σε κρεμότητα, επί των οποίων τελευταίες μέρες μιας που είναι να κάνουμε μια περαιτέρω προσπάθεια βελτίωσης ακριβώς το πνεύμα αγαστής συνεργασίας και να ευχαριστήσω με την ευκαιρία τον ε, κύριο Λίζεκ και τους κοιόδης συζητητές που άλλωστε όπως είναι παράδοση της Επιτροπής μας συνεργάστηκαν Πολύ καλά. Στρατηγική αυτονομία. Λοιπόν, αυτός ο όρος είναι παρόν και έχει παραμείνει και στη δική μου έκθεση. Ίσως ε, θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο, όχι για να αμφισβητήσουμε αυτόν τον όρο, αλλά να το θεωρήσουμε ως μια διαδικασία και όχι ως μια κατάσταση. Είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει και τις σχέσεις μεταξύ Ένωσης και ΝΑΤΟ. Δεν είναι αντιφατικό, με τις σχέσεις αυτές είναι ένα από τα μέσα για τον οποίο η Ευρώπη προχωρεί προς μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε, βλέποντας και τη συμφωνία που φτάσαμε στη δική μου έκθεση, να βρούμε μια θέση παρόμοια. Γιατί νομίζω πως είναι παρόμοια και αυτή η, η θέση. Όσον αφορά τώρα τα βασικά θέματα που συζητάμε τώρα. Ε, ο ρόλος του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να το πούμε αυτά πιο σωστά, αυτό στο πλαίσιο του τομέα ασφάλειας και άμυνας. Νομίζω πως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και δύο πράγματα και νέα. Η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης του Μπαρόζου, που ρητά μίλησε για ευρωπαϊκή πολιτική στο πλαίσιο και στον τομέα των ε, αμυντικών δυνατοτήτων και επίτα χτες προχτές ανακοίνωσε ο Μπαρνιέ μια task force αμυντική. Εγώ νομίζω θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, μια πολιτική διάσταση της έκθεσης πέρα από τα τεχνικά ζητήματα που εξάλλου αφορούν και άλλες επιτροπές όταν θα χρειαστεί να μιλήσουν για το 8ο πρόγραμμα δρά... Ε, πλαίσιο κτλ. Ήτρα κτλ. Εμείς μπορεί να είμαστε θετικοί σε μια ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των και των στρατιωτικών δυνατοτήτων, όμως κατά βάση με δύο ή μάλλον τρεις όρους. Πρώτος είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ει βάρο άλλων πολιτικών. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πρόσθετη η πόρη και όχι αναδίπλωση. Δεν μπορούμε δηλαδή να μειώσουμε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ένα είδος έρευνα υπέρ μια ενό άλλου. Στο 8ο, με συγχωρείτε. Επίτα δεν μπορούμε να δώσουμε τα ευρωπαϊκά χρήματα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας έτσι όπως είναι είτε θα πρέπει να κάνουν σημαντικά βήματα προς τον εξευρωπαϊσμό αυτού του τομέα, την πραγματική δηλαδή οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής άμυνας, είτε ας το ξεχάσουν ότι εμείς με κάποιο τρόπο θα προωθήσουμε και θα δώσουμε κίνητρα για να διατηρηθεί το status quo και άρα θα αντισταθμίσουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτή η ευρωπαϊκή πόρη μπορεί να είναι μόνο ένα, μια βοήθεια. Ε, και τέλος, επιβάλλεται και δημοκρατικό έλεγχο, γιατί από τη στιγμή που έχουμε συναπόφαση Ευρωπαϊκό προπολογισμό με κοινοτική μέθοδο και ούτω καθεξής, είναι σαφέ ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε οποιαδήποτε λογική που να λέει ότι ναι, αλλά αυτό το πράγμα εκεί θα το αποφασίσουν τα εθνικά κράτη για λογαριασμό του. Αυτή είναι η πολιτική θέση λοιπόν. Αυτή τώρα την αυτοσχεδίωσα λίγο για να σα το διατυπώσω αυτό, αλλά ως πολιτικό μήνυμα θα μπορούσε αυτό να ενισχυθεί σε μια συμβιβαστική τροπολογία που να αφορά αυτήν την πτυχή. Τέλος, για το πακέτο. Με εντυπωσιάζει η θέση του συναδέλφου Νικολάη που περίμενα ότι αφού είναι από την Άλτε θα το υπεράσπιζε πιο συνεκτικά ενώ λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για την, άμυνα, για την βιομηχανία άμυνας, θα πρέπει να ισχύσουν εκεί οι κανόνες της ιστορικής αγοράς εκεί και θα ήταν παράδοξο εμείς που το Κοινοβούλιο που ανέκαθεν υποστήριζε την εφαρμογή του φορολογικού πακέτου, να ακολουθήσουμε τις πιο συντηρητικέ θέσει και να πούμε ναι, α διατηρήσουμε τι εξαιρέσει. Α διατηρήσουμε τα συστήματα που έχουμε ένα σωρό μικρέ εθνικές επιχειρήσεις που κάνουν συγκεκριμένα πράγματα για τις δικές τους ε, ένοπλες δυνάμεις και αυτό να εμποδίσει τελικά τη συγκέντρωση, τη μοιρασιά του βάρους και το καθεξής. Γενικά εντάξει είναι, αλλά υπάρχουν με κάποιες φράσεις που ίσως θα έπρεπε να αλλάξουν για να αποφευχθούν οι αμφισημίες. Δηλαδή, στην άμενα και στις θέσεις, γίνονται ε, με μέσα τα οποία ήδη υπάρχουν για τις ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις, δηλαδή Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, ε, η πρόθεση της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης, αλλά όχι μέσω αναχρονιστικών ε, πολιτικών και που γίνονται σε, πολιτικό, σε εθνικό επίπεδο και που δεν μπορούν να ευνοήσουν το συγκεκριμένο τομέα. Πρόκειται για έναν βιομηχανικό τομέα όπως και οι άλλοι και άρα θα πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κινηθούμε. Ίσως λοιπόν να ήταν πολύ γενναιόδωρος ο εισηγητής στη σύνταξη των συμβαστικών τροπολογιών και θα πρέπει λίγο να τις ξαναδούμε. Κύριε Μπουτικόφερ, θέλετε πάλι το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξεπλάγει όταν είπατε ότι δεν ε, πρέπει εδώ να εμπλακούμε σε κομματικές ιδεολογικές ε, αντιπαραθέσεις. Αν μιλάμε όμως για ιδεολογίες θα πρέπει να σας πω με τεκπλήξεως ότι η προοδευτική πλευρά της Επιτροπής ζητά περισσότερο ανταγωνισμό και η δικιά σας πλευρά λιγότερο, πράγμα που με εκπλήσει. Κατά τα άλλα πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν ζητώ περισσότερη συνεργασία και πιο ενισχυμένη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και αν ε, ε, με κατηγορείτε για τέτοια ε, ιδεολογικά πτέσματα η πολιτική μου ομάδα θα γελούσε. Θέλω όμως πελέον των αστείων εδώ να αναφερθώ στο θέμα της στρατηγικής αυτονομίας που θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον και όπως έγινε στην έκθεση καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε μία ενιαία γλώσσα γλώσσα. Όσον αφορά όμως το θέμα το οποίο αναφέρατε ε, για την ε, ε, κατάσταση και απογραφή των αμυντικών μέσων και ότι πρέπει να υπάρξει μία βελτίωση θεωρώ ότι αυτό είναι λαθασμένο διότι μειώνονται οι αμυντικές δαπάνες και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατάσταση για να ζητήσουμε περισσότερο pooling and sharing και αυτά τα οποία έχουμε προσυζήτηση αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκώς φιλόδοξα. Μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερα και αν εγκαταλείψουμε το ε, αμυντικό γραφείο, να, αν αφήσουμε το αμυντικό γραφείο να κάνει ό,τι θέλει, θα είχαν περισσότερες κοινέ ιδέες πέραν της ε, πολιτικής, της εθνικής ανεξαρτησίας στα κράτη-μέλη από ό,τι νομίζετε. Γι' αυτό ε, και αυτή τη στιγμή εφόσον εφόσον ε, ε, ε, θέλουμε να παρουσιάσουμε σαν χριστουγεννιάτικο τραπέζι το, την ευρωπαϊκή έρευνα και να πούμε βάλτε χέρι και εκεί δεν είναι η σωστή πολιτική και γι' αυτό η λύση που ανέφερε ο κύριος Γουαλτιέρη δηλαδή να υπάρξει μία κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση μου φαίνεται συμπαθητικό αλλά δεν αντικατοπτρίζει αυτό που προτείνεται στο κείμενο. Οπότε, γιατί ε, τώρα όταν αναφερόμαστε εις ε, την ε, ευρωπαϊκή αμυντική κατάσταση και δεν είναι το μόνο θέμα, όπως και στο Γαλιλαίο και στο Ίτερ, τα κράτη-μέλη θέλουν να βάλουν χέρι και τους λέμε ε, εάν τα, θέλετε να αναφερθείτε αμυντικό, το, στην αμυντική κατάσταση και προϋπολογισμό μη δώσετε πόρους και τότε δεν μπορεί ε, να υπάρξει χρηματοδότηση για την ε, έρευνα των εξοπλισμών αυτά θα κατανολωθούν κάπου αλλού αυτό θέλουμε δηλαδή δεν θέλουμε να μας δώσουν τα κράτη-μέλη περισσότερα χρήματα αλλά να τους πούμε σας παρακαλώ εμείς ε, Έχουμε ένα προϋπολογισμό αλλά εκεί μπορεί να χρηματοδοτηθούν και ε, το τάλις και άλλα προγράμματα. Λοιπόν, ε, δεν νομίζω ότι είναι η σωστή μέθοδος για να μπορέσει κανείς να έχει επαρκή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Θέλω να σας πω και εγώ μερικά πράγματα στα ρουμανικά, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ αλλά θα παρουσιάσω ρουμάνικα την φιλοσοφία μας. Προσπάθησα να παρουσιάσω μία λύση, γιατί αν θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκές δυνατότητες πρέπει να συνεργαζόμαστε με την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Στις, ε, στην Ανατολική Ευρώπη λέγεται ότι πάντοτε μας δίδουν μία βιομηχανία ήδη μεταχειρισμένων, δεύτερο χέρι και θα θέλαμε και εμείς να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στην αμυντική βιομηχανία. Όλα τα κράτη-μέλη θα, μπορούσαν, θα έπρεπε να μπορούν να αντιδρούν όπως συνάδει με την αμυντική τους πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι ένα είδος έκθεσης αυτό, στο οποίο πάντα κανείς έχει την τάση να θέλει να πετύχει την τελειότητα. Ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπετε έχουμε την τάση να κοιτάμε πολύ μακριά μπροστά στο μέλλον και έχουμε και την φιλοδοξία να ετοιμάζουμε ιδανικά μοντέλα για το μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είχε σαν προσανατολισμό αυτή την συνολική ιδέα, αλλά συγχρόνως θέλαμε να μιλήσουμε και για πράγματα τα οποία είναι φυκτά, τα οποία μπορούμε να πετύχουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήθελα να είμαι και ρεαλιστής στην προσέγγισή μου. Οπότε συμφωνώ με τον κύριο Κόφερ ότι δεν συμπεριλάβαμε δηλαδή πράγματα που έχουν να κάνουν με το ιδανικό μας για το μέλλον. Αυτή είναι μια γενική παρατήρηση που έχω να κάνω. Κατά τα άλλα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για... και για τα θετικά σας και για τα αρνητικά σας σχόλια. Γιατί εδώ είμαστε για να συζητάμε. Αυτή είναι η ουσία της δουλειάς μας. Προκειμένου στη συνέχεια να καταλήγουμε σε συμβιβασμούς. Γι' αυτό και πρότεινα πολλές συμβιβαστικές λύσεις πάνω στις οποίες πρέπει να δουλέψουμε παρετέρω. Έχουμε στην στρατηγική αυτονομία. Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε στις πολιτικές μας ομάδες, εκτός αν το έχουμε ήδη κάνει. Πάντως κύριε Μπουτικόφερ, θέλω να σας πω ότι η χώρα μου, η Πολωνία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τέτοιο πάντα πίστευε ότι πρέπει να έχουμε πολύ στενή συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε, αντίθετα. Άρα λοιπόν με τίποτα δεν ήταν η πρόθεσή μου να προτείνω ότι οι σχέσεις και οι δεσμοί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να αποδυναμωθούν στον ε, τομέα της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Κάθε άλλο. Αν εσείς έτσι ε, καταλάβατε την έκθεσή μου, να ξέρετε ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Κάθε άλλο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας κάθε φορά που αυτό είναι εφικτό. Τώρα, Βαϊμάρη και γενικά το θέμα αυτό. Συμφωνώ και θα ξανακοιτάξω την έκθεση, θα προσπαθήσω να την τροποποιήσω σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά τώρα τις δαπάνες για την έρευνα. Στην άμυνα και στην τεχνολογία άμυνας. Αντιλαμβάνομαι και δεν ήταν πρόθεσή μου να πω ότι η πόρη αυτή, η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να περιοριστεί εξαιτία των περικοπών που κάνουν τα κράτη-μέλη στους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς. Δεν ήταν δικιά μου πρόθεση αυτή και ούτε πιστεύω πως κάποιος από εμά πιστεύει ότι μπορούν να αντικατασταθούν οι πόροι αυτοί. Οι περικοπές στον προπολογισμό είναι μεγάλες αυτές που γίνονται στα διάφορα κράτη-μέλη που δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις εθνικές δαπάνες μέσω της έρευνας. Όχι, δεν ήταν αυτό ως εντύπωση που ήθελα να δώσω. Δεν λέω ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτές τις δαπάνες από τις ερευνητικές. Όχι. Η ομάδα μου πιστεύει ότι πρέπει να μείνει ανοιχτό πάντως ως δυνατότητα και να περιμένουμε. Πρόεδρος εγώ λέω όχι. Είπα ότι να έχουμε λίγες μέρες ακόμα να το συζητήσουμε στις πολιτικές μας ομάδες και να ξανασυναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα. Μα το έχουμε ήδη αποφασίσει για την επόμενη εβδομάδα, αλλά όχι μόνο για αυτή την ιδέα της στρατηγικής, για αυτή την έννοια, γιατί συμφωνούμε με αυτήν. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλετε να αποφύγετε τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ και ότι θέλετε να ενισχυθεί ο ρόλος μας μέσα στο ΝΑΤΟ και τις επιχειρήσεις του. Η έγκριση θα γίνει στις 17 Νοεμβρίου. Η επόμενη εβδομάδα είναι Στρασβούργο, έτσι. Και το Δεκέμβριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Το τελευταίο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα είναι η ετήσια συνέλευση του ΝΑΤΟ 10 Οκτωβρίου 2011 στο, Βουκουρέστι, Βουκουρέστι έλαβε χώρα τη συνέλευση αυτή η ετήσια του ΝΑΤΟ με μεγάλη συμμετοχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπήθηκε από την κυρία Μαντουρέλα, από μένα και τον κύριο Πάσκο. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλα τα θέματα που απασχολούν την Υποβιτροπή μας. Το κύριο θέμα ήταν το Αφγανιστάν, αλλά βέβαια και η Λιβύη. Οι σχέσεις ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και τη νέα στρατηγική μετά τη Λισαβόνα, οι σχέσεις ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετείχαμε ενεργά στη συζήτηση. Πιστεύω ότι ήταν μια καρποφόρα συζήτηση για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Λυπάμαι βέβαια που μόνο τρεις ήμασταν. Ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να συμμετέχει περισσότερο. Αυτά. Τίποτα άλλο. Αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, τότε έληξε η συνεδρίαση της Υποπιτροπής μας για σήμερα. Okay. Listen, listen. I believe Putikoffer doesn't understand anything.